Συνάδελφοι, το επόμενο και τελευταίο σημείο σήμερα διάταξη πριν από τη μεσημερινή διακοπή θα είναι η δήλωση της Επιτροπής αναφορικά με το συντονισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανασυγκρότηση στην ΑΕΤ. Να ζητήσω από την κυρία Γιώργεβα και τον κύριο Πίμπαξ να καθίσουν και να ζητήσω από την κυρία Γιώργεβα να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κύριους και τις κυρίες βουλευτές για την προσοχή που εξακολουθούν να επιδεικνύουν για την ΑΕΤ. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Πίμπαλξ, τον Επιθυνό για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, να σου πω ποιες είναι οι ανθρωπιστικές προκλήσεις και τι κάνει η Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα έχουμε την συνέχεια της ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικά όσον αφορά τη στέγαση, την υγιεινή και την υγεία η μετακίνηση 1,3 εκατομμυρίου αστέγων στο Πόρτο Πρέν σε προσωρινές κατοικίες είναι κάτι το δύσκολο γιατί έχουμε το θέμα της ιδιοκτησίας της γης, της μετακίνησης των συντριμιών και της υγιεινής. Οπότε έχουμε κάπου μεταξύ 10 και 30.000 ατόμων που ζουν σε προσωρινά στρατόπεδα σε περιοχές πλημμυρών και καθώς πλησιάζει η εποχή των τυφώνων θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς και με τη διαχείριση γενικά των στρατοπέδων. Δίνουμε ιδιαίτερη βάση στην συγκέντρωση ήδη εφοδίων που είχαν εξαντληθεί πηγαίνουμε και άλλα εφόδια και βεβαίως ε, πρέπει να υπάρξει και μία οικοδόμηση δυναμικού της αιτανής πολιτικής προστασίας που βγήκε δυνατότερη από την κρίση. Βεβαίως πρέπει να δούμε τις ανάγκες και τον παρακτή βοήθεια εκεί όπου βρίσκονται οι άνθρωποι για να μην έχουμε μαζικές μετακινήσεις. Πρέπει λοιπόν η βοήθειά μας να φτάσει όλη τη χώρα, όχι μόνο στο Πορτοπρέντς, και με αυτό τον τρόπο συνεισφέρουμε στη μείωση της πίεσης που ασκείται στην πρωτεύουσα. Με την ίδια λογική έχουμε μια προσέγγιση για όλη την ίσο είτε αφορά το θέμα των αιτινών προσφύγων, είτε τα ζητήματα επιμελητίας και το πώς θα πάμε εφόδια για την εποχή των ε, θύελων και παίζει σημαντικό ρόλο η Δομινικανή Δημοκρατία, δεν την έχουμε ξεχάσει. Επίσης, ο συντονισμός των δωρητών για να εκμεταλλευτεί ο καθένας το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά εμείς ήμασταν πάντα υπέρ του συντονισμού από τον ΟΗΕ. Και όταν ήμουν στην ΑΕΤ είχα την εντύπωση πως πράγματι αρκετά καλά τα πήγαμε και οι ε, ομάδες πολιτικής προστασίας των χωρών και εμείς. Τέταρτον, να διασφαλίσουμε τη μετάβαση από την ανθρωπιστική βοήθεια στην ανασυγκρότηση. Συνεργαστήκαμε στενά με τον κύριο Πίμπαλξ για να διευκολύνουμε αυτή τη μετάβαση και θα σας δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα στον τομέα των τροφίμων ενθαρρύναμε τις τοπικές αγορές, ακόμα και αν είναι πιο ακριβό, να απευθυνθούμε στους αγρότες, να δημιουργήσουμε ζήτηση για να ανακάμψουν και αυτοί και δεύτερον υποστηρίξαμε προγράμματα μισθωτής εργασίας για να περάσουμε από την βοήθεια στην ανάκαμψη. Τέλος, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στα αποτελέσματα. Η Ευρώπη είναι το νούμερο 1 στον όγκο βοήθειας πρέπει να είναι και νούμερο 1 στα αποτελέσματα και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον αδελφό μου τον κύριο Πίμπαλξ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιέρωσε 1 δισεκατομμύριο 235 εκατομμύρια ε, για την IT και είναι μεγαλύτερος δωρητής παγκοσμίω για την ανασυγκρότηση της IT. Θα είναι η Ένωση συμμετέχει περισσότερο και στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της IT ε, και χαίρομαι γιατί η Ισπανία, η Γαλλία και είχαν απευθύνει την έκκληση αλλά ακόμη και άλλες χώρες όπως η δική μου πατρίδα που δεν είχαν ιδιαίτερες σχέσεις προηγουμένως με την ΑΕΤ αφιέρωσαν σημαντικά κονδύλια από τον Εθνικό Προϋπολογισμό για την υποστήριξη της χώρας αυτής. Η συνδιάσκεψη των δωρητών ε, είχε πολύ αίσια έκβαση η κυβέρνηση της ΑΕΤΙΣ ε, ανέλαβε την ε, ιδιοκτησία σε αυτό το σχέδιο. Δεν είναι ότι έμεινα μέτοχη σε όλες αυτές τις προσπάθειες ανασυγκρότησης. Είχαμε σημαντική συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά προβλέψαμε και κάποιους μεταβατικούς ε, μηχανισμούς συντονισμού υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού της ΑΕΤΙΣ και της κυρίας Χιλαρή Κλίντον και θα, θα φροντίσουμε ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα κονδύλια και να μην χαθεί τίποτα. Ε, τώρα προτεραιότητά μας, προτεραιότητα, μας είναι να δρομολογήσουμε την βοήθεια το συντομότερο δυνατό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ετοιμάζουν τη νέα στρατηγική με πρόγραμμα υποστήριξη της ΑΕΤ. Θα ενισχύσουμε την, ε, τις διαδικασίες για την ε, οικοδόμηση του οίκου της Ευρώπης στην ΑΕΤ για να διευκολύνουμε τις εργασίες και μάλιστα θα πάω αυτή τη βδομάδα στην ΑΕΤ για να παράσχω και την απτή υποστήριξη στην ε, βοήθεια που χρειάζονται οι υποδομές αλλά και τα θέματα της διακυβέρνησης. Χρειαζόμαστε πέντε χρηματοοικονομικές συμφωνίες για συνολικό ποσό πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ και θα εγκαινιαστούν και κάποια έργα όπως αποκατάσταση του δικού δικτύου μεταξύ του ακροτηρίου της ΑΕΤΙΣ και του Πόρτο Πράνς, που βρίσκει φυσικά σύμφωνα την κυβέρνηση, αλλά θα βοηθήσει και την προσέγγιση μας για κάλυψη ολόκληρης της νήσου. Θα ενισχυθούν και η το ικανότητα διακυβέρνησης. Υπάρχει και η σχολή της Μιραμπέλ και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, όπως ζήτησε και ο πρόεδρος ΑΕΤΗΣ. Επίσης, θα φροντίσουμε ότι η δημοσιονομική ενίσχυση θα φτάνει το συντομότερο δυνατό. Και αυτή δεν είναι τυφλή ενίσχυση, δεν είναι επιταγή που δίνεται εν λευκό. Έγιναν πολλές επιτόπιες επισκέψεις και θα σας, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα κονδύλια. Επίσης, θα έχουμε τακτικές ενισχύσεις για την επίβλεψη της διαδικασίας ανασυγκρότησης και θα κρατώ συνεχώς ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο που σημειώνεται στην ανασυγκρότηση της ΑΕΤ. Δεν θα είμαι μόνο βέβαια εγώ, αλλά όλο, ολόκληρη η Επιτροπή. Η Κρυσταλίνα, η Πατεκπρόσωπο, Βαρονιάστον, αλλά και άλλοι επίτροποι θα μεταβούν στην ΑΕΤ για να βοηθήσουν την ανασυγκρότηση. Και ο Επίτροπος Μπαρνιέ έχει μεταβεί στην ΑΕΤ. Οπότε το θέμα τη ανασυγκρότησης ΑΕΤ δεν είναι αρμοδιότητα ενό και μόνο επιτρόπου, αλλά του συλλογικού οργάνου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση θα πρέπει να εξετάσουμε τρόπου για τη βελτίωση τη παροχή συνδρομή. Γιατί δεν θα πρέπει η ΑΕΤ να παλινδρομήσει σε μια κατάσταση σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την προσφορά της παγκόσμιας κοινότητας και να βρούμε τους τρόπους που θα υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο γιατί τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν οι αρχές της ΑΕΤ και ο λαός της ΑΕΤ. Και δύο πτυχές φαίνονται κυρίως. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πτυχή, θα πρέπει να, έχουν, να, να υπάρχουν στενές επαφές μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αλλά και ολόκληρης κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ε, παναϊτιανή συμφωνία σε ό,τι αφορά το το πρόγραμμα ανασυγκρότηση. Από οικονομική άποψη, το μακροοικονομικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στη Νέα Υόρκη, στη διάσκεψη των δωρητών, θα πρέπει να είναι αυστηρό και να επικεντρωθεί στα θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος της ανισότητας, της αδικίας και της φτώχειας. Ευχαριστώ. I Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα θα ακούσουμε τους εκπροσώπους ε, των πολιτικών ομάδων. Πρώτα εκ μέρους του ΕΛΚ για δύο λεπτά ο κύριος Μίτσελ. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους. Τρία σημεία θα ήθελα να φέρω πρώτα απ' όλα η μέθοδος και τα μέτρα μέτρησης των αναγκών ανοικοδόμησης. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε πως ε, θα εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας και τρίτον βεβαίως δικαιώματα ιδιοκτησίας και το πόσο ευάλωτοι είναι άνθρωποι που ζουν σε καλύβες πάνω σε γη που δεν τους ανήκει. Πρώτα απ' όλα, για την ανοικοδόμηση. Πήγα πρόσφατα στη διάσκεψη της Παγκόσμιας ε, Τράπεζας για το έγγραφο το οποίο είχαμε ένα εγχειρίδιο δηλαδή και βεβαίως ε, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η έκθεση υπάρχει Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το βιβλίο. Δεύτερον, όσον αφορά τις δεσμεύσεις μας, χαίρομαι ιδιαίτερα για τα 207 εκατομμύρια. Θα τα δώσουμε θα, ή θα ξανάρθουμε σε ένα χρόνο και σε, ένα, ή σε πέντε χρόνια και θα λέμε τα ίδια. Θα δώσουμε επιτέλους αυτά τα λεφτά σε μια φτωχή χώρα την οποία δεν μπορούμε να την αφήσουμε μόνη της. Τρίτον, η έκταση της καταστροφής ήταν τέτοια ώστε πρέπει να δούμε και τη ζημιά και το γιατί ήταν τόσο εκτεταμένοι. Οι άνθρωποι ζούσαν σε ρεματιές, στην άκρη των βουνών σε καλύβες γιατί δεν είχαν ιδιοκτησία. Αν είχαν δικαιώματα ιδιοκτησίας θα έχτιζαν κανονικά σπίτια που θα είχαν κάποια ελπίδα να αντισταθούν σε ένα σεισμό. Σκεφτείτε το αυτό. Και πάλι κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ, η κυρία Κρετού τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. μισή λεπτό. Η κατάσταση πόρο απέχει από το να σταθεροποιηθεί, όπως είπαν και οι δύο επίτροποι. Τα ίδια αναφέρουν και οι μη ανθρωπιστικές, ε, κυβερνητικές οργανώσεις που βρίσκονται επί τόπου και δρούν. Χρειάζεται να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Είναι ιδιαίτερα κατεπήγον το ζήτημα διότι η περίοδος των βροχών επίκειται και οι υποδομές, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τις ε, μεταφορές, είναι σε ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση. Είναι προφανές ότι νέα προβλήματα θα προκύψουν αργότερα σε επίπεδο υποδομών, στέγασης ε, του πληθυσμού κλπ. Χρειαζόμαστε λοιπόν να προωθήσουμε το ζήτημα της ε, ανοικοδόμησης και της ανασυγκρότησης ορφανά ή και παιδιά τα οποία έχουν διαχωριστεί από τις οικογένειές τους βρίσκονται σε ιδιαίτερα επισφαλή κατάσταση ως εκ τούτου χρειάζεται να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την ανθρωπιστική πτυχή της κρίσης ε, στην ΑΕΤ διότι υπήρξαν προβλήματα με τις ε, υιοθεσίε των ε, παιδιών της ΑΕΤ. Χαίρομαι που η ο συντονισμό τη Ευρωπαϊκή Βοήθεια και τη Ανασυγκρότηση στην ΑΕΤ αποτελεί μία από τι προτεραιότητε ε, τη Κομισιόν. Ο κ. Γκέρντ έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ε, επίκειται η περίοδο των ε, καταιγίδων και των θυελών στην ΑΕΤ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε αύξηση της τις βοήθειας. Απαιτούνται λοιπόν παράλληλα να υπάρξει και μια βοήθεια στην παντεποδομή. Η οικοδόμηση των καταστρεμμένων κατοικιών χρειάζεται χρόνο και εξάλλου η, αντιμετώπιση των μελλοντικών προβλημάτων που θα προκύψουν από ενδεχόμενη θύελα ή πλημμύρε ε, θα είναι πολύ σημαντικέ. Χρειάζεται λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθειες, ε, χρειάζεται παράλληλα να προωθήσουμε την βοήθεια προς την οικονομία για να βρούνε δουλειά οι άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους. Χρειάζεται μια δημοσιονομική ενίσχυση της ΑΕΤ, βράχη πρόθεσμα, καθώς επίσης και η δέσμευση για την αποκέντρωση. Η διάσκεψη των δωρητών που διεξήχθη στην Ηνωμένα Έθνη 31 Μαρτίου αποτέλεσε επιτυχία. Το τι θα παραμείνει αυτή την διάσκεψη όταν θα έχουν όλα ξεχαστεί, εκτός από τις ε, ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ανάγκη ε, πρόθεση της οικονομίας, ε, κάτι το οποίο αναφέρει και ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αναφέρεται σε μια ανάγκη αύξησης της τάξης του 8% την επόμενη πενταετία. Επίσης η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είναι η κατεξοχήν οικονομική προτεραιότητα. Σήμερα η ΑΕΤ έχει ανάγκη από το 80% των εσόδων της από τις για να χρηματοδοτήσει τα γεωργικά προϊόντα. Τρίτον, ε, σχετικά με τα κριτήρια της ε, αποτελεσματικότητας, της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας πρέπει να αξιολογήσουμε την ανάπτυξη να είτε. Επίσης, για να ενταχθεί η ανάπτυξη στον, ε, στη διάρκεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ανάπτυξη των, του κοινωνικού τομέα είναι σημαντική. Θα πρέπει επίσης ε, να λάβουμε υπόψη ε, και την ε, βοήθεια η οποία χορηγείται και τι περιμένουμε για να υλοποιήσουμε στην πράξη την έκθεση του Μισελ Μπαρνία. Και τέλος η συμβόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση προβλήματος της ΑΕΤ ήταν πολύ σημαντική. Ευχαριστώ τον Ινίπατο αρμοστή των Επιτρόπων Επιτρόπους και Αντιορτζίεβα. Ευχαριστώ κύριε Γκόρεν, ο κύριο Τσαρνέσκι έχει το λόγο. Ένα λεπτό για τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Θα ήθελα εκ μέρους πολιτικής μου ομάδας, αλλά και εκ μέρους του συντονιστή της ομάδας μας, του κυρίου Ντέβα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η σημερινή ενίσχυση προς την ΑΕΤ είναι τριπλάσια από ό,τι περίμενε η κυβέρνηση της ΑΕΤ αρχικά. Και μάλιστα η βοήθεια αυτή ανέρχεται σε 1,5 περίπου δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί Αρχικά ήταν πολύ λιγότερο το ποσό που αναμένατε και μέσα στα, επόμενα 2,5 χρόνια μπορεί να έλθει και σε 4 δισεκατομμύρια συνολικά ευρώ η συνολική ενίσχυση προς την ΑΕΤ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και όπως έλεγε ο κύριος ε, Ντέβα συντονιστής, είναι πολύ σημαντικό το θέμα του ελέγχου δρομολόγηση αυτής της βοήθειας, γιατί είναι πολύ αδύναμη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της ΑΕΤ. Και κυκλοφορούν διάφορες αμφίβολε αμφίβολες εντυμότητες ελίτ στην ΑΕΤ. Καλό θα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξει αν πραγματικά τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στα σωστά χέρια και πώς ναι. αξιοποιούνται. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει εκ μέρους της ΓΚΟ ο κύριος Λιαρίκ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι υποσχέσεις δωρεών στη συνδιάσκεψη των δωρητών να λάβουν σάρκα και οστά, να μετατραπούν σε απτά κονδύλια και να φτάσουν πραγματικά στους ε, παραλήπτες αυτά τα κονδύλια. Δεν αρκεί όμως αυτό για να ανασυγκροτήσουμε ε, με αηφόρο τρόπο την ΑΕΤ. Γιατί πολλά οφείλουμε στο λαό της ΑΕΤ και θα πρέπει να τον βοηθήσουμε. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε μεγάλη γενεοδορία και αλληλεγγύη. Ελοχεύει όμως ο κίνδυνος να ξεχάσουμε την τραγωδία που βιώνουν ή αιτινοί, τα αδέρφια μας οι αιτινοί. Γιατί όπως είπατε είναι κατεπίγουσα η κατάσταση και επιτακτική ανάγκη να δώσουμε βοήθεια. Γιατί ε, θα πρέπει ε, να χτιστούν αμέσως νοσοκομεία, ε, οικίες, σχολεία, ενώ οι πλημμύρες καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση, θα πρέπει να γίνει καλύτερο συντονισμό της κατανομής ε, της ανθρωπιστικής και επιστηστικής βοήθειας ε, και της υγειονομικής φροντίδας και επίσης να εξασφαλίσουμε μια υφόρο γεωργική ανάκαμψη της ΑΕΤ για να μην εξαρτάται από γεωργικές εισαγωγές. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Αιτινών. Όλες οι κρατικές ε, προμήθειες και όλοι οι διαγωνισμοί ε, ανασυγκρότησης θα πρέπει να είναι διαφανείς και να περιλαμβάνουν ρήτρες για την απασχόληση, την στέγαση, την υγεία κτλ. Γιατί σωστή ανασυγκρότηση δεν πρόκειται να γίνει αν δεν στηριχθούμε στον ίδιο το λαό και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους ε, συλλόγους και τα σωματεία των γεωργών. Θέλουμε ένα νέο σχέδιο και όραμα για την IT που θα αποκλείει τη φτώχεια, την εξάρτηση και την υπερίσχυση των οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η απογύμνωση των Αιτινών δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του φρικτοφτούσισμού σεισμού, αλλά και της κυριαρχίας πολλών άλλων ξένων δυνάμεων προς τη χώρα αυτή. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον Αιτινό λαό να ανακτήσει την πολιτική και οικονομική του κυριαρχία. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπέλτερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά την καταστροφή έγινε μια αξιολόγηση για τις προτεραιότητες και κατέληξαν οι ΜΚΟ όπως δεν γίνεται χρήση της ε, τοπικής εμπειρίας που υπάρχει για να βοηθηθεί ο πληθυσμός. Θα έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ο τοπικός πληθυσμός στην ανοικοδόμηση και καλό θα είναι και οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ να έρθουν σε επαφή με τον τόπιο πληθυσμό και εσείς να σκεφτείτε προς αυτή την κατεύθυνση, να βοηθεί από μόνη της η ΑΕΤ. Κάτι άλλο. Τα τρόφιμα που στέλνουν είπα, και οι λοιπές χώρες καλή ιδέα μοιάζουν, αλλά τι συμβαίνει, καταστρέφεται έτσι η γεωργία της ΑΕΤ και 50% πλέον εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια και 50% της οδειάς της IT πηγαίνει χαμένη. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτεί και η Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση γιατί χρειάζεται πάρα πολύ θάρρος για να δείτε την κατάσταση κατάματα. Τα βασικά λοιπόν, στέγαση, εκπαίδευση, αυτά και εύχομαι καλή επιτυχία στην Κομισιόν πάνω από όλα εδώ πέρα σας. Now, next speaker is Mr. Σας ευχαριστώ. κύριος Μάουρο για να το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, στάση των Επιτρόπων. Πραγματικά ε, έγιναν πολλά πράγματα μπορώ να πω ότι φυσικά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ούτε να αρκεστούμε. Ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα είναι απαραίτητο δεδομένων των, της κατάσταση κατάστασης που επικρατεί στην χώρα. Το ζήτημα της έκτακτης ανάγκης ε, ίσως να μην έχει ακόμα καταλήξει. Συνεχίζουν ε, οι άνθρωποι να πεθαίνουν από την πείνα, την ε, την δίψα κλπ λίγο θα χρειαστούν να αντιμετωπίσουν την περίοδο των κυκλώνων και των βροχών. Τι χρειάζεται, όπως είπε ο Επίτροπος, υπάρχει συντονισμό ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και να συνδυαστεί με μια πιο αποτελεσματική σχέση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδιαίτερα με αυτές που δρούν επί τόπου και είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις ανάγκες των πολιτών και να φροντίσουν να υπάρξει συμμετοχή των πολιτών στην ανοικοδόμηση και την συγκρότηση. Όλοι λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε πως ε, το να αποτελούμε σημείο αναφοράς για την ΑΕΤ και για τους πολίτες ε, σημαίνει ότι πρέπει να τους ε, καταδείξουμε ότι θα πρέπει να αποκτήσουν εκ νέου την αξιοπρέπειά τους, δηλαδή να έχουν μια ελπίδα ευτυχίας και ευημερία μετά από αυτόν τον τραγικό και τρομερό σεισμό που τους έπληξε. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γιερέρο, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε και κύριοι Επίτροποι. Τα πρώτα λόγια μου είναι, αφορούν ευχαριστίες αλλά και τα συλληπιτήρια τα οποία απευθύνονται προς τους τέσσερις Ισπανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στην ΑΕΤ. Ήταν απεσταλμένοι, ε, εξειδικευμένοι ε, αλλά ε, απεστάλησαν ως μέλη μιας ανθρωπιστικής αντιπροσωπείας και το ελικόπτερό τους δυστυχώς κατέπεσε και συνετρίβει. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση τις περισσότερες φορές ανάμεσα στην ασφάλεια και την ε, ανθρωπιστική δράση. Του εναντίον, ε, δίχως την ασφάλεια είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την ε, ανεξαρτησία και την ουδετερότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε στις στρατιωτικές δυνάμεις πολλών κρατών μεταξύ αυτών και της Ισπανίας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ΑΕΤ μας ε, αποδεικνύει ότι η φτώχεια αυξάνει ε, το αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών και η έλλειψη διακυβέρνησης ε, αποτελεί τροχοπέδι για τη δυνατότητα μιας αποτελεσματικής απάντησης. Συνήθως η ένδια και η έλλειψη διακυβέρνησης προχωρούν χέρι-χέρι και αυτό συνέβη και στην ΑΕΤ. Επίσης, αντί να υποστηρίξουν τις διαδικασίες οικοδόμησης, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη διακυβέρνηση της ΑΕΤ, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο που είχαμε θέσει στη Νέα Υόρκη, ότι δηλαδή η ΑΕΤ θα πρέπει να είναι αυτή η οποία θα κατευθύνει την αντιδεκρότησή τη και η κοινωνία των πολιτών η οποία θα συμμετέχει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Γκερέρο. Ο κύριος Μισελ, συγγνώμη. Ε, θα ήθελα να συγχάρω τους δύο επιτρόπους ε, που είναι αρμόδιοι για τα ζητήματα αυτά και για τις παρεμβάσεις τους που ε, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικέ. Ο σεισμό της Αϊτή μας έδειξε την ε, αδελφοσύνη αλλά και την αλληλεγγύη. Θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ τις προσπάθειες και το κουράγιο των πληθυσμού της ε, Αιτή, τη διασπορά της Αϊτή, ε, των δωρητών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Οι θεσμικές δυναμίες στην Αϊτή είναι γνωστές και αυτή η καταστροφή απέδειξε το εύρος, το τραγικό, την τραγική έκταση στην ε, Νέα Υόρκη στην διάσκεψη καταδείχθη ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να υποστηρίξει, να υποβοηθήσει το πρόγραμμα της ΑΕΤΙΣ. Η θα πρέπει λοιπόν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά η βοήθεια των δωρητών θα πρέπει να τύχει ικανού συντονισμού και όπως είπε ο πρόεδρος να πετύχει την ε, αποτελεσματική ανασυγκρότηση και την ε, μέσω της σύστασης μιας ε, προσωρινής επιτροπής αλλά και τη δημιουργία ενός καταπιστεύματος επίσης να ενισχύσει τη διακυβέρνηση των θεσμών που θα στηρίζονται στην, στο δίκαιο και ελπίζω η ανασυγκρότηση και η ανοικοδόμηση, κύριε Επίτροπη, να, να, να πάρει στον δρόμο, κάτι το οποίο, για το οποίο κανείς δεν αμφιβάλλει. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Στίφλερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατοντάδε χιλιάδες άνθρωποι μένουν ακόμη σε καταβλισμούς, ενώ έχει αρχίσει η εποχή των βροχών και πλησιάζει και η εποχή των τυφώνων και ελλείψη σημαντικού δυναμικού και κρατικής ικανότητας, η ανθρωπιστική βοήθεια αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών να παράσχουμε με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια. Ήμουν στη Νέα Υόρκη στις 31 παρελθόντος Μαρτίου στη συνδιάσκεψη των δωρητών και ε, χαίρομαι για την προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ενός δισεκατομμυρίου 300 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη τριετία για την ανασυγκρότηση της ΑΕΤΙΣ και επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποφάνθηκε με νέα φωνή αυτή της είπα της εκπροσώπου κυρίας Άστον. Η διεθνή κοινότητα κάνει ό,τι μπορεί, αλλά θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να χρησιμοποιηθούν σωστά, αποτελεσματικά και θα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή των μεθόδων και μέτρων εφαρμογή, γιατί φυσικά ο αιτινός λαός θα πρέπει να είναι αυτός που θα, ε, θα λάβει τη βοήθεια. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την γεωργική παραγωγή της ΑΕΤ και να βοηθήσουμε την ανάκαψη της γεωργίας. Θα πρέπει φυσικά να χρησιμοποιηθούν, να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για την ανασυγκρότηση της ΑΕΤ και να σκεφτούμε επιτέλους ε, για την ίδρυση της δύναμης πολιτικής προστασίας που την αναμένουμε εδώ και καιρό. Ο κύριος Αρσένης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επίτροποι. Η ανθρωπιστική κρίση στην ΑΕΤ ανέδειξε και δυστυχώς αναδεικνύει ακόμη τα προβλήματα των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών Αντιμετώπισης Διεθνών Ανθρωπιστικών Κρίσεων. Πρέπει να δημιουργήσουμε πάγιους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Ακόμη δεν έχουμε ουσιαστικά πάγια κονδύλια στον ευρωπαϊκό προπολογισμό για την οικονομική αρρωγή σε τρίτε χώρε και η βοήθεια στην αϊτή δόθηκε κυρίω σε διμερέ επίπεδο από ευρωπαϊκέ χώρε. πρέπει η βοήθεια να φτάνει άμεσα. ακόμη και μετά από μια εβδομάδα η βοήθεια δεν είχε φτάσει στου ανθρώπου που χτυπήθηκαν από το σεισμό στην ΑΕΤ. πρέπει οι ευρωπαϊκοί πόροι να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. χρειαζόμαστε να έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό που να μπορεί να σχεδιάσει να υλοποιήσει γρήγορα και αποτελεσματικά προγράμματα ανθρωπιστική βοήθεια. προφανώ η καταστροφή στην αϊτή προήλθε από ένα σεισμό όμω αντίστοιχε ανθρωπιστικέ κρίσει μπορούν κάλλιστα να προκληθούν και από άλλα καιρικά φαινόμενα όπω τυφώνε τροπικέ καταιγίδε πλημμύρε ξηρασίε φαινόμενα που εν ώψη των κλιματικών αλλαγών θα αυξηθούν σημαντικά σε συχνότητα και σε ένταση. αγαπητοί συνάδελφοι όπω γνωρίζουμε καλά η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο που εμεί οι χώρε προκαλέσαμε αλλά πολλές φορές είναι οι φτωχέ χώρες που πληρώνουν τις επιπτώσεις. έχουμε ένα κλιματικό χρέος προς τις ευάλωτες χώρες και πρέπει να μάθουμε τις αδυναμίες μας στην αντιμετώπιση της κρίσης στην αϊτή για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ε, παγκόσμιες υποχρεώσεις μας στο μέλλον. ευχαριστώ πολύ. Κύρια Γεωργίευα και κύριε Πίπαλξ, μετά την φοβερή τραγωδία, την καταστροφή της ΑΕΤΙΣ, πρέπει να δούμε και το μέλλον. Η διάσκεψη στη Νέα Υόρκη πριν από δύο εβδομάδες απέφερε 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποσχέσεις. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία είχε σχεδιάσει η Ιταλία και η ΑΕΤ υποσχέθηκε 1,2 δισεκατομμύρια η Ευρώπη και το θέμα είναι τώρα πώς θα σταθεροποιηθεί η νήσος και είναι μακρά η διαδικασία. Το ερώτημά μου προς εσάς τους δύο είναι πώς αξιολογείται το σχέδιο δράσης της αιτινής ε, κυβέρνησης και πώς θα φροντίσετε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά αυτά τα μέσα για να πάρει στον πληθυσμό που τα χρειάζεται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και πώς μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε με το 1,3 εκατομμύρια άστεγους και πώς θα φροντίσουμε μέσω πρόθεσμα να υπάρξει μια κατασκευή υποδομών στην ΑΕΤ. Βεβαίως είναι οι άμεσα πληγέντες που μας ενδιαφέρουν, αλλά καλά θα κάνουμε να δούμε τι θα γίνει και με την πολιτική σταθερότητα στην Ίσο. Το κράτος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύθραυστο. Ο πληθυσμός θεωρεί πως δεν πηγαίνει βοήθεια εκεί που χρειάζεται και τι μπορούμε να κάνουμε για την πολιτική κατάσταση στην Νήσο και για να βοηθήσουμε την προσέγγιση της ε, κυβέρνησης. Υπάρχει τώρα μία ενδιάμεση επιτροπή ανάκαμψης της Ε, έχετε ένα λεπτό και μιλάτε ήδη δύο λεπτά, λέει ο πρόεδρος. Για τον Δε Κλίντον θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ε, σκοπεύετε να κάνετε για αυτό το θέμα και για την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ Κύριε Κατσμάρ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στρίφλερ για αυτά που μας είπε και τους δύο επιτρόπους για τις δηλώσεις τους. Νομίζω ότι πολλά, πολλές από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά μας ε, βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση. Έχουμε δύο φάσεις ανασυγκρότησης, δεν το είπαμε αρκετά. Έχουμε καταρχήν τη μέσο και μάσο, μακροπρόθεσμη βοήθεια εξόδου από την κρίση, γιατί αυτή τη βοήθεια χρειάζονται οι φτωχότεροι κάτοικοι της ΑΕΤ. Μίλησε η κυρία Γεωργίευα. Και η δεύτερη φάση είναι η ανασυγκρότηση, η ανοικοδόμηση, που θα πρέπει να είναι φόρος και χρειάζεται να εφαρμοστεί συντονισμός. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η ιδιοκτησία αυτού του σχεδίου ανασυγκρότηση θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την Αιτινή κυβέρνηση και τον Αιτινό λαό. Οι Αιτινοί ίδιοι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ανασυγκρότησής τους. Επίσης, εμείς τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο συντονισμένη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι που ασχολούνται και με το θέμα αυτό οι δύο επίτροποι. Σας ευχαριστώ κύριο Ζουβά για ένα λεπτό. Πρόεδρε, η Ευρώπη συνέβαλε με εκατομμύρια ευρώ, με σκηνές, με στρατιώτες, τρόφιμα κλπ. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο δήμαρχος του Πόρο Πρένς που τον Φεβρουάριο χρησιμοποίησε τον όρο καταστροφή. Όχι για να φέρει τα αποτελέσματα του σεισμού, της συνέπειά του, αλλά για την απόλυτη αποδιοργάνωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και αυτό είναι ερώτημα που πρέπει να θέσουμε σε αυτούς μας. Πώς θα αποφύγουμε λοιπόν αυτή την αποδιοργάνωση η οποία κόστησε πάρα πολύ στην ΑΕΤ. Σε αυτό το ερώτημα, Πρόεδρε, κυρία και κύριε Επίτροπε, υπάρχει μια απάντηση, την γνωρίζουμε όλοι. Αναφέρθηκε η σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας. Πότε η Κομισιόν προτίθεται να υποβάλει επιτέλους στο Κοινοβούλιο την σύσταση ενός τέτοιου οργάνων τέτοιου σώματος ε, συμπεριλαμβανομένων μέσων ε, μεταφοράς κλπ. Μπορούμε να το πράξουμε άμεσα πριν από την επόμενη καταστροφή. Παρακαλώ πάφτε να μιλάτε για συντονισμό, απλώς πράξτε τον, υλοποιήστε τον. Ευχαριστώ κύριο Σιλβέστρης για ένα λεπτό. Αξιότιμοι συνάδελφοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπω τα αποτελέσματα της διάσκεψης των δωρητών, διότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά πολύ πιο σημαντική ήταν και ε, ο τρόπος ε, για τον οποίο αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι. Η ΑΕΤ θα πρέπει να εξέλθει πιο δυνατή από ό,τι στο παρελθόν πριν δηλαδή την πλήξη ο, το σεισμός δεν θα πρέπει να αποκαταστήσουμε απλά τις πόλεις που υπήρχαν. Πρέπει να οικοδομηθούν σωστά κτίρια, αλλά γι' αυτό χρειάζονται χρήματα. Χρειάζεται επίσης και τα τεράστια μέσα τα οποία διαθέτουν οι διάφοροι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί να υλοποιηθούν σωστά με τον κατάλληλο συντονισμό. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν, αφού εδώ ε, κατακρίναμε κάποιες καθυστερήσεις αρχικές ε, όπου η Ευρώπη με, δεν μπόρεσε να ε, καταστεί αποτελεσματική ευθύς εξ αρχής. Σήμερα χαιρετίζουμε την εξαιρετική εργασία που κάνουν τα θεσμικά μας όργανα, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι αυτή η γραμμή θα συνεχιστεί μέσω ενός μακροχρόνιου προγράμματος και με την παρουσία των θεσμικών μας οργάνων θα υλοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιλβέστρες. Τώρα έχουμε τη διαδικασία Κάτσου Διάη. Κυρία Ζαρμπόσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Επιτέλους δρομολογείται η διεθνής βοήθεια προς την ε, ΑΙΤ. Εκτός από Καναδούς στρατιώτες έδωσαν το παρόν στην ΑΙΤ και Σλοβάκοι στρατιώτες. Και η Σλοβακία ήταν μία από τις χώρες που έδρασαν ε, αμέσως για την παροχή ενίσχυσης, γιατί δεν ήταν πολλές οι χώρες που έσπευσαν να βοηθήσουν την ΑΙΤ. Μπορούμε τώρα να διαπιστώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήχε ανθρωπιστική βοήθεια και υλική βοήθεια προς την ΑΕΤ, αλλά χωρίς και την επιστημιστική βοήθεια, χωρίς είδωρ, χωρίς μηχανήματα, δεν θα ήταν αρκετά αποτελεσματική αυτή η βοήθεια. Δεν χρειάζεται μόνο καλή βούληση, αλλά χρειάζονται και εφόδια και πρακτικοί τρόποι χρήση αυτή τη βοήθεια. Γι' αυτό και είμαι υπέρ τη ε, πρόταση για την ανάγκη καλύτερου συντονισμού τη ε, Παγκόσμια ανθρωπιστικής βοήθεια, όπω είπαμε και στο ψήφισμά μα για την ΑΕΤ. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην υποστήριξη τη παιδεία ε, και να ενισχύσουμε του μηχανισμού αντίδρασης σε τέτοιου είδου θεομηνίε. Η επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Φραντσέσκα Κέλλερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ αγαπητοί επίτροποι για την παρουσίασή σας και για τις προσπάθειές σας. Συμφωνώ πως καλό είναι να δούμε ολόκληρη την Ίσα. Μπορεί να μην συμφωνώ με αυτά τα οποία λέτε για την προσέγγιση για όλη την Ένωση, αλλά συμφωνώ με την προσέγγιση ολόκληρη την Ίσο. Για τις δε μελλοντικέ ε, δεσμεύσεις πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας γιατί βλέπουμε πως δεν τηρούμε το 0,7 ως κράτη-μέλη. Πρέπει να φροντίσετε εσείς να συμμορφωθούν εδώ τα κράτη-μέλη. Και η πρόοδος στην ΑΕΤ δεν πρέπει να ξεπεραστεί από άλλες πολιτικές που θα μας εμποδίσουν να λάβουμε μέτρα. Πρέπει να υπάρχει πολιτική συνοχής για να μην έχουμε επιτυχία στην ΑΕΤ και μετά όλα αυτά να ερημώσουν λόγω άλλων πολιτικών. Ευχαριστώ και καλή τύχη. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Γετεμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε την IT. Και αυτό είναι σωστό. Αλλά η καταστροφή αυτή κατέδειξε πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει να βελτιωθούν τα της πολιτικής προστασίας. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να αντιδρά γρήγορα σε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να μπορεί να στέλνει ανθρώπους επιτόπου και να βοηθάει τον κόσμο άμεσα και όχι αφού περάσει χρόνος. Σημαντική και αυτή η βοήθεια, αλλά σημασία έχει και η άμεση βοήθεια που δεν την έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε δύναμη ταχεία Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κάποιο άλλο θέλει τον λόγο. Όχι, οπότε θα δώσω τον λόγο στην κυρία Γεωργίευα για να απαντήσει σε ερωτήσει. Ένα... Ευχαριστώ. Και θα αφήσω και λίγο χρόνο για τον κύριο Πίμπαλξ με την άδειά σας. Ήταν χρήσιμη και ενθαρρυντική συζήτηση. Πριν ε, περάσω τώρα στα ερωτήματα αυτά, θα ήθελα όπως και ο κύριος Γκερέρο να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις, τέσσερις, ε, στις οικογένειες των τεσσάρων Ισπανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν και τη συμπαραστασή μου σε όλες τις ομάδες ανασυγκρότησης στην ΑΕΤ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα μεγαλύτερα ζητήματα της πολιτικής. Δηλαδή, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιώσει την αντίδρασή της. Χάρηκα που είδα τον κύριο Μπαρνιέ εδώ εντός σα γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα οπότε θα έχουμε την ευκαιρία στις 26 Μαρτίου στην Επιτροπή Ανάπτυξης να συζητήσουμε πιο λεπτομερώς το πρόγραμμα εργασίας το οποίο συμπεριλαμβάνει για το 2010 την ενίσχυση των δυνατοτήτων ε, ε, της Ένωσης και τη σχετική ανακοίνωση. Και αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ομάδα μας. Θα συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη, με το Κοινοβούλιο για να βρούμε μια λύση η οποία θα βελτιώσει τη δυνατότητα αντίδρασης στις καταστροφές και είναι απλή η λογική εδώ πέρα. Σε έναν καιρό που αυξάνεται η ένταση των καταστροφών και ο προϋπολογισμό μας ε, θα είναι σφιχτός για χρόνια δεν μπορούμε παρά να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό συντονισμό και να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που θα μπορούν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά και εδώ πέρα λέω αποτελεσματικά και όσον αφορά τα αποτελέσματα και όσον αφορά το κόστος. Και θα έχουμε και μια επίσκεψη στη χώρα. Είναι λοιπόν υψηλή προτεραιότητα για την ομάδα μας αυτό τους επόμενους μήνες. Να αναφερθώ τώρα σε τέσσερις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα τον συνδυασμό των άμεσων αναγκών με τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εάν περάσουμε και φύγουμε και αφήσουμε τους ανθρώπους ξεκρέμαστους θα υπάρχουν τραγωδίες και πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα της παροχής τροφίμων. Η κυβέρνηση της ΑΕΤΙΣ πρότεινε να φύγουμε από την παροχή τροφίμων στο να περάσουμε στο θέμα της μισθωτής εργασίας και τρόφιμα έναντι εργασίας. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό παντού ταυτόχρονα και είναι κάτι που παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά όσον αφορά γενικότερα το ζήτημα της διατροφικής ασφαλείας η νέα μας πολιτική στην Ένωση είναι πολύ προοδευτική γιατί τονίζει τσέτερης πάρυμπους. Θα λέγαμε το να ενθαρρύνουμε την παραγωγή επιτόπου όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτό θα συζητηθεί, συζητήθηκε και σε μια πρωινή συζήτηση με αιτινές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και χάρηκα για το ότι και οι ευρωπαϊκές μήκυο έθεσαν αυτό το ζήτημα της διατροφικής ασφάλειας της ΑΕΤΙΣ και της παραγωγικότητας της αϊτινής γεωργίας. Κατόπιν να αναφερθώ στο ζήτημα της στέγασης. Δεν είναι δευτερεύον. Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μετακινηθούν. Για διάφορους λόγους ακόμα και αν είναι ασφαλή τα σπίτια τους, φοβούνται να ξαναμπούνε γιατί υπάρχει τραυματική εμπειρία. Δεύτερον, είναι, έχουν ε, διαμορφώσει γειτονιές και υπάρχει ένας κοινωνικός ιστός. Δεν είναι λοιπόν ε, μόνο απροθυμία, είναι και κοινωνικό το ζήτημα που ακολουθεί μια τέτοια καταστροφή. Και δεν είναι τόσο εύκολο να μετακινηθούν οι άνθρωποι από περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες να πάνε σε πιο ασφαλείς. Αλλά είναι προτεραιότητά μας αυτό το ζήτημα και θα ήθελα να τελειώσω με το θέμα της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και της κυσέως και της οικολογικής. Εγώ δυστυχώς πέταξα πάνω από την Αϊτή και πάνω από τη Χιλή σε δύο εβδομάδες. Πάνω από την Αϊτή είναι μια, η Αϊτή είναι μια κατεστραμμένη νήσος και βεβαίως στην Χιλή η κυβέρνηση επί δεκαετίες κάνει αναδάσωση, σταθεροποιεί το έδαφος και άρα δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον. Κάτι το οποίο βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και έτσι μακροπρόθεσμα πρέπει να σκεφτόμαστε και κάτι άλλο που δεν είναι δικό μου, αλλά επειδή δούλευα στην Παγκόσμια Τράπεζα, συμφωνώ μαζί σας. Αυτό το οποίο προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα για τον συντονισμό, για ένα καταπίστευμα και όσον αφορά τη διαχείριση των έργων, είναι κάτι που πρέπει να το ασπαστούμε. Και εδώ πέρα θα δώσω λόγο συνάδελφο. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι να ευχηθώ μάλλον ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο στο Κοινοβούλιο για να μπορώ να απαντώ. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά θα αναφερθώ σε ορισμένες εξ αυτών. Νομίζω ότι για μας ως Επιτροπή ε, είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική η υποστήριξή σας. Αυτό είναι, αυτό ένα θέμα που αφορά το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, ε, το θέμα της ε, ανασυγκρότησης τώρα. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει μέχρι τώρα είναι η αξιολόγηση, το προγραμματισμό, συζήτησαμε το θέμα με τις ε, μη κυβερνικέ οργανώσεις ε, και φροντίζουμε να συντονίσουμε την όλη διαδικασία και δεν δημιουργούμε κάτι το παράλληλο, απλά μέσω συνεργασίας φροντίζουμε να προχωρήσουμε συγχρόνως ε, και ομαδικά έχουμε αναλάβει κάποιες πολιτικές δεσμεύσεις και νομίζω ότι αυτές θα τις στηρίσουμε και θα τις υλοποιήσουμε. Τώρα, σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, έχουμε ένα, ένα κτηματολόγιο το οποίο φροντίζουμε να ε, γίνει σεβαστό χρειάζεται παράλληλα να προχωρήσει και η πολιτική διαδικασία στην χώρα και να πιστέψει ο λαός σε αυτήν. Αυτή είναι μεγάλη πρόκληση. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε τις αιτιανούς, την κοινωνία τους, προκειμένου να καταστεί επιτυχές. Τώρα, σε ό,τι φορά τη διαφάνεια της διαδικασίας, ε, υπάρχει ένα σύνολο δωρητών φροντίζουμε να υπάρχει η κατάλληλη διαφάνεια και σας διαβεβαιώ ότι τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν όχι μόνο για τους συγκεκριμένους στόχους αλλά και ε, μέσω μιας χρηστής διαχείρισης. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα πρέπει να πούμε ότι όσοι βρουν επιτόπους ε, από τη διεθνή κοινότητα, την ευρωπαϊκή κοινότητα κλπ ε, δρούν αποτελεσματικά και να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου στις οικογένειες των τεσσάρων στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά όλοι όσοι εργάζονται επί τόπου καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να πετύχουν το καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα συνάδελφοι η συζήτηση ολοκληρώθηκε και θα επαναληφθεί στις 15.00. Καλή σας όρεξη.